Ο κύριο Φατούτσο για την έκθεση Μπέλντερ και ένα λεπτό υπενθυμίζω αυστηρά. Signora Presidente, grazie. Eh, Con grande piacere prendo la parola. Με μεγάλη ευχαρίστηση παίρνω το λόγο σε αυτή την τόσο σημαντική κοινοβουλευτική ε, σύνοδο όπου έχουν έρθει εκπρόσωποι και των 27 κρατών μελών. Κάτι το οποίο μου συμβαίνει σπάνια. Ποτέ δεν έχω τόσους πολλούς ακροατές. Και θα πρέπει να εξηγήσω γιατί υπερψήφισα την έκθεση ε, της, του της, ε, του κυρίου Μπάστιαν Μπέλτερ για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τα Δυτικά Βαλκάνια. Εγώ είμαι υπέρ της διευκόλυνσης ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της προσχώρησης των χωρών αυτών στην Ένωση. Θα Πιστεύω ότι οι οικονομικές ε, ενισχύσεις θα πρέπει να είναι πιο σημαντικές από αυτέ που έχουν χορηγηθεί μέχρι τώρα. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να αυξηθούν οι επικοινωνίε με τις, ε, ανάμεσα στην Ευρώπη και στα Δυτικά Βαλκάνια, να προωθήσουμε τον τουρισμό και όλοι οι Βαλκάνοι, είτε είναι νέοι είτε είναι συνταξιούχοι, να ζουν καλύτερα από ό,τι ζούσαν μέχρι τώρα. Ωραία, περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Μαγκίνες. Ο κύριος Μπακού, ένα λεπτό. Πού είναι? Κύριε Μπακό. Whatever. Il n'est pas là, M. Bacot. Ah, ah, c'est 783. Ah, bon, je donne la parole. Λοιπόν, δίνω το λόγο στην κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να καταγραφεί το γεγονός ότι στην έκθεση της κυρίας Μαγκίνες πάτησαν λάθος κουμπί. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την έκθεση της κυρίας ε, Μαγκίνες για την ε, γεωρική πολιτική και την επιστηστική ασφάλεια. Ε, θα, το, έρθω σε επαφή με τις ε, κατάλληλες τεχνικές υπηρεσίες. Εγώ πιστεύω ότι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον. Ναι μεν ε, την σταθερότητα δεν μπορούμε να την εξασφαλίσουμε, αλλά μια κάποια ασφάλεια μπορούμε. Θα πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση των συνεπειών, κυρίως όσον αφορά την, ε, ε, την, την, τη συνέπεια πολιτικής στην επιστηστική ασφάλεια. Και για την ασφάλεια των φυτών, αν δείτε, χρειαζόμαστε μια λεπτομερή ε, αξιολόγηση των συνεπειών και την επιστηστική ασφάλεια θα πρέπει να αντιλαμβάνουμε υπόψη μας όταν κάνουμε αυτές τις εκτιμήσεις. Ωραία. Η κυρία Μαγκίνες για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, γιατί υποστήριξαν την έκθεση και πραγματικά Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό αντικατοπτρίζεται η θέληση και η άποψη του Κοινοβουλίου και των πολιτών της Ευρώπης ε, για τα θέματα αυτά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι θα πρέπει να επανεστιάσουμε στην γεωργική πολιτική ξανά, μέσα στα, κυρίως όσον αφορά τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς ε, που δεν μπορούν να παράγουν τρόφιμα επιτόπου. Αυτό το δισεκατομμύριο της Ευρώπης θα βοηθήσει Όντω Όντως πιστεύω ότι η έκθεση αυτή αποτελεί ένα πρότυπο για το μέλλον, για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την γεωργία και πώ η επιστημιστική ασφάλεια δεν πρέπει να φύγει από την ημερήσια διάταξη. 13.000 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα από την πείνα, από την ασυτεία στον κόσμο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο κύριος Σάνμπεργκ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να εξηγήσω γιατί απήχα από την έκθεση Μαγκίνες. Ε, εστιάζει η έκθεση αυτή σε μια πάρα πολύ σημαντική ε, πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε τρόφιμα σε αυτούς που πεινούν ή σε αυτούς που δεν μπορούν να προμηθευτούν κανονικά τα τρόφιμα. Προφανώ κανείς δεν θα ήταν αντίθετο σε κάτι τέτοιο και δεν είμαι κι εγώ αντίθετο στο πρόβλημα, όμως με την έκθεση είναι ότι εξετάζεται και εξετάζει την κοινή γεωργική πολιτική μεν, αλλά δεν ασχολείται με το γεγονός ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη να μεταρρυθμιστεί και να μεταρρυθμιστεί εκ νέου αυτή η πολιτική δεν, είναι, δεν εξυπηρετεί το καλό των πολιτών, των καλών των αγροτών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης και αν δεν ε, ε, λάβουμε υπόψη μας ε, τις επιπτώσεις στον Ευρωπαίο φορολογούμενο, τα πράγματα δεν θα είναι σωστό. Πιστεύω δηλαδή ότι η έκθεση αυτή δεν ασχολείται με το ουσιαστικό πρόβλημα. Ο κύριος Σεκάσκι, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα περισσότερα τα οποία περιέχονται στην έκθεση Μαγκίνας. Γιατί ξέρετε ότι όλο ένα και περισσότερο τώρα θα ε, αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων στην παγκόσμια αγορά, το οποίο θα έχει όλο ένα και περισσότερες αρνητικές συνέπειες και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτοί που πλήσονται τελικά είναι αυτοί που έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα, αυτοί οι οποίοι τα περισσότερα χρήματά τους θα εξοδεύουν για φαγητό. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο και κυρίως στις ανεψόμενε χώρες αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση πορείας και έτσι να λάβουμε υπόψη αυτά τα προβλήματα της διατροφικής ασφάλειας. Και επίσης θα πρέπει να προσέξουμε και να δούμε πώς δεν θα έχουμε κάποια ε, συστήματα τα οποία φρενάρουν την αγορά τα οποία φρενάρουν τις ενισχύσει στη Γεωργία. Επομένως είναι πάρα πολύ σωστή ιδέα, ιδέα να υπάρξει μια διεθνής εποπτεία των ε, τιμών των τροφίμων και με αυτή την ε, εποπτεία να ελέγξουν τις εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα. Ε, οπότε βέβαια θα πρέπει να βρούμε και ένα σύστημα αποθήκευσης, αποθεματοποίησης τροφίμων σε διεθνή κλίμακα. Ο επόμενος, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, με αυτή την ευκαιρία να σας εξηγήσω γιατί απέσχον όσον αφορά την ε, ψηφοφορία της έκθεσης. Όλο το πολιτικό φάσμα συμφωνεί ότι η διατροφική ασφάλεια είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν συμφωνούμε στον ορισμό αυτής της ενίας. Πολλοί εξημών θεωρούν ότι αυτό σημαίνει έχει εξασφαλιστεί φαγητό για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο παντού, παντού στην ε, ε, οι Άλλοι θεωρούνται μια δικαιολογία για προστατευτισμό. Και μόνο ό,τι παράγεται στην Ευρώπη είναι για τους ε, Ευρωπαίους ε, και πολλοί επικαλούνται τη χαμηλή παραγωγή δεν θα πρέπει να έχουμε πρόφαση την διατροφική ασφάλεια για να φράξουμε τις εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο γιατί πολλές φτωχές χώρες έτσι βρίσκονται σε κατάσταση ε, προβληματική και κάποιοι φτωχοί γεωργοί ε, έτσι καταδικαζούνται σε παινία. Αυτό επομένω ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καταλήλω. Ο κύριο Χίτον χάρη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα συνάδελφο. Εγώ επίσης απέσχον και επί την γραμμή της παραταξής μας αλλά Ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η διτροφική ασφάλεια και σωστά το εδώ στο Κοινοβούλιο στη δε έκθεσή αναφέρθηκε και πιστεύω ότι ψηφίστηκε αυτό το πρόβλημα το οποίο εμείς το δημιουργούμε. Το δημιουργούμε όταν ε, εγκρίνουμε τέτοιες οδηγίες. Ψήφιζουμε μια έκθεση και τρία λεπτά μετά πάμε και ψηφίζουμε κάποια μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την συρρήγνωση της παραγωγής. Αυτό θα πρέπει να το καταγγείλω. Κυρία Ντόιλ, τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μια από τις κύριες ανησυχίες, Πρόεδρε, και ένα από τα κύρια θέματα ω προς την, τα κλειδιά θα έλεγα για την προστασία των τροφίμων, ε, την ασφάλεια των τροφίμων θα ήταν η εξασφάλιση παραγωγή και ασφάλεια σε τρόφιμα στο λεγόμενο αναπτυξόμενο κόσμο όπω και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μην έχουμε ανταγωνιστική σχέση ο ένας προς τον άλλο στην παγκόσμια αγορά με την αύξηση των τιμών για εκείνε τι περιοχέ που δεν έχουν κλιματολογικέ συνθήκε, ή έδαφο κατάλληλο για την παραγωγή τροφίμων και να μην έχουμε και πλεονάσματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τη δική μας παραγωγή ώστε και περιβαλλοντικά αλλά και σε επίπεδο παγκοσμιοποίησης να έχουμε υπεύθυνη στάση ως προς την παραγωγή τροφίμων. Ευχαριστώ κύριε Μπακού. Πρόεδρε, υπερψήφισα την ε, πρόταση για την έκθεση σχετική με την κοινή αγωγή και την ασφάλεια στο τρόφιμα, διότι ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που πολλές φορές έχω επισημάνει εδώ, δηλαδή το κόστος της παραγωγής, την αυξανόμενη παραγωγικότητα και την ε, ιδιαίτερη πτυτικότητα των αγορών τροφίμων, ιδιαίτερα όταν περιορίζονται τα αποθέματα σε τρόφιμα ή μειώνεται η παραγωγή. Εξάλλου γνωρίζουμε πόσο οι πολίτες μας αποδίδουν σημασία όλο και περισσότερη στη γεωργική παραγωγή, στην ποιότητα των τροφίμων ε, και στην κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να δώσουμε τα μέσα αυτά που θα επιτρέψουν την ε, παραγωγή ασφαλών και σε επαρκείς ποσότητες τροφίμων. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τα νέα κράτη-μέλη, χωρίς να υποχρεώνονται να ε, υφίστανται ε, συνθήκες και όρους νομοθεσία η οποία επιδεινώνει την κατάσταση της παραγωγής τους. Για την έκθεση της κυρίας Γκραμπόρσκα παρακαλώ. Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Εδώ βεβαίως έχουμε να κάνουμε με το επίκεντρο, με, το, με το πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα για να πείσουμε, το, για να πείσουμε το, την κοινή γνώμη να υπερψηφίσει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο πολίτης όμως, ιδιαίτερα ο πολιτή στην δημοκρατία της Ιρλανδική Δημοκρατία, κατέστησε σαφές το τι θέλει, ότι δεν θέλει δηλαδή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Άλλωστε και στι προηγούμενε εκλογέ από την κυβέρνηση των εργατικών είχε δοθεί σχετική υπόσχεση και μάλιστα είχε δοθεί και στο παρελθόν αρνητική ψήφο προ την Ευρωπαϊκή Ένωση από του Ιρλανδού πολίτε. Πρέπει να το ακούσει πια αυτό, να το εισακούσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουν περισσότερο έλεγχο από τι Βρυξέλλε και το Στρασβούργο οι πολίτε τη Ευρώπη. Θέλουν τη δική του κυβέρνηση. Ο καθένα θέλει το δικό του νομοθετικό σώμα να λαμβάνει τι αποφάσει που τον εκφράζουν και που τον εκπροσωπούν. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, διαρκώ θα διοχετεύουμε τα χρήματα του φορολογούμενου σε μια προσπάθεια να πείσουμε τον πολίτη όταν προσέχεται στι κάλπε να αλλάζει γνώμη. Δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη ο πολίτη. Χάρκιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να σημειώσω ότι πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση, πρόταση. Θέλουμε πάντοτε βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρχεται πιο κοντά στου πολίτε και αυτό δεν μπορούμε να το καταφέρουμε εάν δεν συμβάλλει ο πολίτη. Γιατί υπάρχουν δύο τύποι δημοκρατία. Μία που έχουμε εδώ, η εκπροσωπευτική, και η άλλη είναι συμμετοχική. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να επιτυχούμε με τη συγκεκριμένη έκθεση. Όμω ο διάλογο μέσα στι κοινωνίε με τον πολίτη είναι αμφίδρομο. Πρέπει να ακούμε δηλαδή αυτά που έχει να πει ο πολίτη και πρέπει αυτά που έχει να πει ο πολίτη να τα εισακούν οι θεσμοί, τα θεσμικά τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν το 1,5 εκατομμύριο για τη συμμετοχή ε, μπορεί να επηρεάσει, μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Δεν συμφωνώ φυσικά με το προλαλήσαντα γιατί πιστεύω όντως ότι η συνθήκη της Λασαβόνα εάν τη θέση ισχύ θα μας επιτρέψει να, να συνεργαστούμε με τον πολίτη, να τον φέρουμε κοντά στην Ευρώπη σε πιο ουσιαστικό και συμμετοχικό τρόπο. Ελπίζω λοιπόν να τεθεί σε, συνθήκη, σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας αφού εγκριθεί, αφού κυρωθεί μάλλον από τους υπόλοιπου. Κύριος Αχάναν. Πολλά θα μπορούσαμε να εξάγουμε από τον τίτλο ε, της, ε, του κειμένου αυτού «Προοπτικές ανάπτυξης του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας». Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν εφαρμόζεται. Τρεις, ε, τρεις φορές ε, το, την αρνήθηκαν οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Ιρλανδοί και με σημαντικά ποσοστά. Δεν ξέρω αν είναι ο οργολικός ο τίτλος «Προοπτικές ανάπτυξης ε, του διαλόγου». Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ε, δεν ξέρω αν, ότι οι πολίτες μπορούν να καταλάβουν τον ίδιο τρόπο τις λέξεις αυτές ε, όπως εμείς, δηλαδή να δημιουργηθεί μια κάποια προπαγάνδα για να προωθήσουμε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Ο διάλογος εκ των πραγμάτων ε, συνεπάγεται δύο μέρη τα οποία, διαλόγου, τα οποία διαλέγονται μεταξύ τους. Ε, λοιπόν, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εξάγει τα συμπεράσματά της. Κύριος Καμάλ, ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε την δυνατότητα να εξηγήσω την ψήφο μου. Όταν διάβασα τον τίτλο προοπτικές ανάπτυξη του διαλόγου των πολιτών στο πλαίσιο τη συνθήκη τη Λισαβόνα θυμήθηκα κάτι που είχε πει ο Μαχάτ Μαγκάντι για την δυτικό πολιτισμό που είπε καλή ιδέα. Λοιπόν, το ίδιο στα ίδια σκέφτομαι το διάλογο των πολιτών μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Όντω, καλή ιδέα. Αν είχαμε έναν διάλογο των πολιτών, αν είχαμε μια αμφίδρομη συζήτηση. όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητή, η συζήτηση, ο διάλογος, χρειάζεται δύο μέρη. Όμω, μήπω θα έπρεπε καταρχάς να δούμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας τι λέει. Μονάχα ένας οργανισμός ε, υπάρχει για να προωθεί αυτή τη ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Πόσες οργανώσεις ε, που είναι αντίθετες στη συνθήκη, στη συνθήκη της Λισαβόνας θα χρηματοδοτηθούν και θα προωθηθούν. Γι' αυτό οι πολίτες της... Οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν του εδόθη η ευκαιρία, απέρριψαν τη συνθήκη τη Λισαβόνα για την έκθεση Γκερέιρο, κύριο Καμάλ. Για την έκθεση Γκερέρο, κύριε Καμάλ. Can you just remind me what it was on? Sorry. Uh, oh, it's on fisheries. Yeah. Α, για την αλία. Ναι, ναι, να σας πω σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή που επιδείξατε, συνάδελφοι πάρα πολύ συναντοπαστικέ όλε αυτέ τι ψηφοφορίε που έγιναν σήμερα. Ένα ώρα θα μπορούσα να σα πω γι' αυτό. Λέμε ναι στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αλληλευτική πολιτική. Όμω έχουμε φτάσει σε αντιφατικό σημείο. Γιατί αν θέλουμε βιώσιμη αλληλευτική πολιτική, τότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα δικαιώματα τη κυριότητα, τι γίνεται με λύσει τη αγορά θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια δικαιώματα τα οποία να επιδέχονται θέσει εμπορία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ε, κληροδότησή του από τη μία φουρνιά στην άλλη, να μην έχουμε επομένω ε, μεθόδου ε, ιονί κομμουνιστικέ, κεντροκατευθυνόμενε. Έτσι θα προστατεύσουμε και του αλληλευτικού πόρου και τελικά όλοι θα την πληρώσουμε. Τώρα θα γίνει μια διακοπή, λέει ο Πρόεδρο. θα διακοπεί η συνεδρία και θα συνεχίσουμε μετά τι εξηγήσει ψήφου, μετά από αυτή την πανηγυρική συνεδρία που θα αρχίσει τώρα.